Πρέπει να σας κάνω μερικές ανακοινώσεις. Πρώτον, θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 226 εδάφιο 4 του κανονισμού μας δεν υπήρξε αίτημα να υποβληθεί σε ψηφοφορία το διορθωτικό που έγινε χτες στις 5 το απόγευμα. Οπότε θεωρείται εγκεκριμένη αυτή η πρόταση. Δεύτερη ανακοίνωση σε σχέση με τις δύο συστάσεις αποφάσεων από πλευράς ε, της Επιτροπής